την ε, Τετάρτη μαζί με τον πρόεδρο του Συμβουλίου θα υπογράψω πέντε εκτελεστικές πράξεις δυνάμει του άρθρου 78 του κανονισμού και θα εγγραφούν στα πρακτικά της παρούσας